των ε, κρατών. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους από Ήτρε, ΕΚΟΝ και από την, στις μεταφορές και την ΡΕΓΙ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλες τις επιτροπές Έμπλιτρε και έκον και τώρα ο υποψήφιος μπορεί να ε, προβεί σε μια καταληκτική ε, δήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είναι η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να ξανασκεφτώ το ζήτημα του πακέτου των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου, θα ήθελα να ξανασυζητήσουμε τις προτεραιότητες της κάθε επιτροπής του καθένα Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του πακέτου επενδύσεων και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα ο κοινοτικός προϋπολογισμός και ποια χρηματοοικονομικά μέσα θα θέλατε και μέτρα θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε περισσότερο. Επίσης, εάν με εγκρίνετε, θα ήθελα τη βοήθειά σας για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, ε, ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά. Ε, πολλά κράτη αντιτάχθηκαν, αλλά τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα για πιο φιλόδοξες ε, προσπάθειες για να δημιουργήσουμε μία πραγματικά ενιαία αγορά, να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να προωθήσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους όπως σας είπα και πριν, θα ήθελα να καταβάλω προσπάθειες για πραγματικές επενδύσεις και πραγματική συνεργασία. Ε, παρόλο που δεν είμαι πολιτικός ε, πλέον, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ ζητημάτων και αξιών αλλά πολλές φορές οι πολίτες, ε, ε, στους πολίτες δεν γινόμαστε αρεστοί όταν δίνουμε μάχες ως πολιτικοί. Γιατί να μην επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα θέματα που μας βρίσκουν σύμφωνος. Δυστυχώς δεν έχει επανέλθει η εμπιστοσύνη στους πολίτες στον κοινό μέσο άνθρωπο. Δεν θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να βρούμε τα ζητήματα που μπορούν να μας βρουν σύμφωνους και όπου δεν υπάρχει διαφωνία και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και αυτό το πνεύμα συνεργασίας για να προωθήσουμε τις επενδύσεις, ε, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για αυτή την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Μιλώ γρήγορα πολλές φορές, γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους και το Προεδρείο καθώς και τη Γραμματεία για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να εκφράσω τις απόψεις μου. Ευχαριστούμε κύριε υποψήφιε ε, επίτροπε. Θα ήθελα ο κύριος Γκουαλτιέρη να λάβει το λόγο για ορισμένα τελικά σχόλια. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον υποψήφιο επίτροπο Κατάινεν για την ενδιαφέρουσα ακρόαση, τα μέλη της ΕΚΟΝ καθώς και την ΙΤΡΕ. Ε, Θα ήθελα τα μέλη της ε, ΕΚΟΝ να μεταβούν στην ακρόαση του κυρίου Χιλ. Δίνω το λόγο στη Μαρίτα Ουλσκόπ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις σας και τον κύριο Κατάινεν ιδιαίτερα για τις απαντήσεις του. Περάσατε δύσκολες ώρες, αλλά νομίζω ότι έτσι έχει η διαδικασία των ακροάσεων και φτάνουμε και στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ακρόαση αυτή και δεν είναι και η τελευταία να το τονίσω αυτό. Ευχαριστώ τους συμπροέδρους και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τα μέλη του ε, Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα ορισμένες ε, πληροφορίες στις 2.30 έχουμε την ακρόαση του κυρίου Τίμερμανς, υποψηφίου αντιπροέδρου. Επίσης διάσκεψη των ε, προέδρων που είναι ανοιχτή σε όλους. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες. Επίσης, στη Νιάμι, οι συντονιστές της ΙΤΡΕ Econ Employment, στις 6, στις 6 αυτό. Και στις 7 συνεδρίαση με την ΕΜΒΗ. Ευχαριστώ και την κοινή γνώμη που μας παρακολουθεί και βρίσκεται κοντά μας. Σας ευχαριστώ όλους.